Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνουμε εδώ τη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 11.30 το πρωί. Θα συζητήσουμε τώρα ένα άλλο σημείο στις σημερινή διάταξη, στην έκθεση της κυρίας Νίκης Τζαβέλα, τον ενεργειακό χαρτί πορείας για το 2050. Έχει το λόγο η συγκεκριά για 4 λεπτά καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλανε σε αυτή την έκθεση και κυρίως τους σκιώδεις εισηγητές τη γραμματεία και τους πολιτικούς συμβούλους. οι βασικοί πυλώνες μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού η διαφοροποίηση των προμηθευτών και πηγών ενέργειας οι ανταγωνιστικές τιμές και η ενεργειακή αποδοτικότητα αυτές οι πολιτικές συμπληρώνονται από τον γενικό στόχο της μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Κυρίες και κύριοι, στην τοποθέτησή μου αυτή θα ήθελα να μιλήσω πάνω και πέρα από αυτά που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω έχοντας κατά νου την ευθύνη που φέρουμε όλοι εδώ μέσα ως νομοθέτες για την επιβίωση, διαβίωση και καλοζωία των ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με την ενέργεια. κυρίες και κύριοι ας μιλήσουμε λοιπόν για την ενέργεια και να κάνω κάποιες προτάσεις για την ενεργειακή μας πολιτική που απαιτούν ρεαλισμό μετριοπάθεια υπέρβαση επίγνωση της πραγματικότητας και συμβιβαστικό πνεύμα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία ενέργειας και περιβάλλοντος. Δογματικές προσεγγίσεις και από τις δύο πλευρές έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργειακή φτώχεια των Ευρωπαίων πολιτών και την αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Ως Ευρωπαίοι χάσαμε το αγωνιστικό δημιουργικό πνεύμα μας καταργώντας μορφές ενέργειας. Αντί να τις βελτιώσουμε και να τις κάνουμε φιλικές προς το περιβάλλον. Η Ευρώπη κυρίες και κύριοι χτίστηκε από θαραλέους άντρες και γυναίκες που αντιμετώπισαν τα πάντα ως πρόκληση και όχι ως απειλή. Όταν στοχεύεις σε ένα καλύτερο μέλλον δεν καταργείς. Δημιουργείς το καλύτερο με αυτά που έχεις. Στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη πάνω από 50% του οικογενειακού προϋπολογισμού πάνε για το κόστος της ενέργειας. Πού θα πάει αυτό. Στη Βουλγαρία βγήκανε στους δρόμους, έπεσε η κυβέρνηση εξαιτίας του κόστους της κυβέρνησης, της ενέργειας. Δεν θέλω να είμαι Κασάνδρα, αλλά προβλέπω μια αλυσίδα κοινωνικών αντιδράσεων εξαιτίας της ενεργειακής φτώχειας και σε αυτή την έκθεση την οποία συζητάμε ήταν καλό που από την πλευρά των σοσιαλιστών για πρώτη φορά μπήκε και η κοινωνική διάσταση της ενέργειας. κύριε επίτροπε επιδείξτε μια γενναία στάση για την αξιοποίηση του σχιστολιθικού αερίου. το οφείλετε στους λαούς της ευρώπης. κύριε επίτροπε γνωρίζω ότι έχετε πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας των κοιτασμάτων της νοτιοανατολικής μεσογείου. στηρίξτε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των κοιτασμάτων αυτών δημιουργώντας επιτροπή ενέργειας της νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής μεσογείου με μόνιμα μέλη την ελλάδα την κύπρο την ιταλία και την ευρωπαϊκή ένωση. άλλωστε αυτό το δικαίωμα σας δίνει το άρθρο 194 της συνθήκης της Λισαβόνα, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση δικαιούται να λαμβάνει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Μπορείτε να ορίσετε την Ελλάδα σε ένα περιφερειακό κέντρο που θα συγκεντρώνει και θα μεταπολεί φυσικό αέριο και όπου θα διαπραγματεύονται και θα καθορίζονται οι τιμές φυσικού αερίου για την περιοχή έτσι θα αποκτήσουμε ως ευρωπαίοι ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά φυσικού αερίου που αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβη για τα κράτη μέλη. η ευρώπη πρέπει επιτέλους να δείξει εμπιστοσύνη στις ενδογενείς πηγές ενέργειας που διαθέτει είτε είναι ορυκτά καύσιμα ή ο άνεμος του βορρά ή ο ήλιος του νότου. αν δεν αναγνωρίζαμε το ρόλο των ανανεώσιμων πηγών δεν θα ήμασταν αντικειμενικοί. έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν αλλά δεν μπορούμε να ζητούμε δεσμευτικούς στόχους την ώρα που δεν υπάρχει κεντρική ευρωπαϊκή διαχείριση στα ενεργειακά. η μετάβαση δηλαδή στις ανανεώσιμες πηγές δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. ευχαριστώ πολύ. E, ο επόμενος ομιλητής είναι ο Επίτροπος. Ο κύριος Öttinger. Κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές, εμείς ε, θέλαμε τελικά να ξεκινήσουμε μία συζήτηση η οποία μας οδηγεί στις επόμενες δεκαετίες η οποία μας δείχνει την κατεύθυνση πώς θα δώσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σε αυτή την πολιτική ενέργειας η οποία θα είναι και βιώσιμη. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει άλλο τομέα εκτό από αυτών τη ενέργεια που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε μία στρατηγική ε, ένα στρατηγικό σχεδιασμό βασισμένο στην ασφάλεια. Και βεβαίως εδώ αναφερόμαστε στην ασφάλεια όσον αφορά την, τις πηγές ε, προμήθειας και αυτό και στην ενέργεια που προέρχεται από τον άνθρακα, από τα άλλα από τις άλλες ε, πηγές, αλλά και από την γεωροθερμία και από τις νέες πηγές ενέργειας. Και αυτό βεβαίως σημαίνει και υποδομή, σημαίνει και τα δίκτυα, σημαίνει την απόδοση, την υψηλότερη απόδοση και φυσικά εδώ ο σχεδιασμός δεν μπορεί να περιοριστεί σε 5-10 χρόνια όπως σε άλλους τομείς όπου χρειάζονται 3 ή 5 χρόνια αλλά παραδείγματο χάρη για τον εξοπλισμό μηχανημάτων χρειάζεται 8 με 10 σχέδια, ε, χρόνια σχεδιασμός για τα αυτοκίνητα βλέπουμε ότι ο χρόνος είναι πολύ πιο περιορισμένος από ότι στον τομέα της ενέργειας, όπου εδώ ο σχεδιασμός ξεπερνάει τα 15, 20, 30 χρόνια. Αυτά σας τα λέω, γιατί πραγματικά, όπως είπατε κύριε Τόμας, εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε το σχεδιασμό στο μέλλον, την ασφάλεια. Και η τεχνολογία όπως αναφέρατε στην Γαλλία για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι τεχνολογία προ 40 ετών. Μιλήσατε για τις αδειοδοτήσεις και βλέπετε ότι σήμερα ζητούνται επεκτάσεις αυτών των αδειών για 40, 50, 60 χρόνια. Και το 2020 θα φτάσει πριν το καταλάβουμε. Και καταλαβαίνετε ότι οι επενδύσεις που πρέπει σήμερα να σχεδιαστούν δεν έχουν γίνει στο βαθμό που έπρεπε. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις. Και για το 2030, 40, 50 είναι οι στόχοι μας όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα αυτών. Και εδώ βεβαίως έχουμε διαφορετικά σενάρια. Και αναφέρονται εδώ τρεις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Επενδύσεις ε, στις υποδομές για το τομέα της ενέργειας, κάτι το οποίο βεβαίως είναι πλεονέκτημα και σε καμία περίπτωση αρνητικό στοιχείο, όπως παρουσιάζεται πολλές φορές. Μας δίνει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από μειονεκτήματα όσον αφορά τη βελτίωση της απόδοσης ε, της ενέργειας αυτό είναι σαφώς και ενδιαφεσβήτητα ένα σωστός δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα επικοδομητικά σας ε, σχόλια και πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να ξαναδούμε τις συστάσεις αυτής της έκθεσης. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί στόχοι. Και με το 2020 Εάν δεν το πετύχουμε αυτό, θα οδηγηθούμε σε ένα κατακαιρματισμένο μέλλον στο τομέα της ενέργειας και βλέπουμε ότι η πράσινη βίβλος που έχει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει την βάση αυτών των στόχων και αυτής της πολιτικής. Η μείωση των εκπομπών του διοξείδου του άνθρακα το ερώτημα αν αρκεί αυτός ο στόχος για τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό βεβαίως. Αλλά, αλλά, παρόλα αυτά, είμαι υπέρ παράλληλων στόχων ρεαλιστικών που θα βασίζεται στην μείωση των εκπομπών, θα βασίζεται όμως και σε μια ρεαλιστική πολιτική για καλύτερη απόδοση της ενέργειας. Και αν κοιτάξει κανείς τους στόχους όπως θέσαμε το 2007, βλέπουμε ότι υπήρχε ομοφωνία στο Συμβούλιο. Όλα τα κράτη-μέλη υποστήριξαν αυτούς τους στόχους. Και το άρθρο 149 και όσο αυτό το άρθρο ισχύει, δίνει τις αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Και ξέρετε ότι σήμερα η επιλογή των κρατών μελών υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας παραμένει αρμοδιότητα των κρατών. Και αν 20 κράτη-μέλη δεν θέσουν ένα κοινό στόχο για τις ανανεώσιμες παραδείγματος χάρη πηγές ενέργειας, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω λοιπόν εκ των προτέρων ότι βλέπουμε το κλίμα να αλλάζει, να επηρεάζεται από αυτή τη δραστηριότητα. Και έχω τη φιλοδοξία μαζί με εσάς να προετοιμάσουμε επικοδομητικές προτάσεις για την επόμενη δεκαετία και για τις επιλογές της επόμενης δεκαετίας. κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι δημιουργικό. Και αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πού θέλουμε να πάμε όσον αφορά τις επιλογές μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θεωρώ ότι σήμερα θα πρέπει να στοχεύσουμε το 10% όπως έχει σήμερα η κατάσταση αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους, παραδείγματος χάρη την μελλοντική παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και όσον αφορά παραδείγματο χάρη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020 ο στόχος είναι 32%. Κάτι το οποίο βεβαίως ε, αν θέλουμε να υλοποιηθεί, χρειάζεται τις προσπάθειες, τις αποτελεσματικές προσπάθειες όλων μας. Τώρα, όσον αφορά την προμήθεια και τις πηγές προμήθειας, θα ήθελα να πω ότι η, το το φυσικό αέριο από το σχιστόλιθους είναι κάτι το οποίο όπως βλέπετε θα μπορούσε να αποτελέσει κάποιες άλλες δυνατότητες. Σήμερα εξαρτώμαστε από τις χώρες που έχουν ε, πετρέλαιο. Τις χώρες στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη. Και βλέπουμε ότι σήμερα οι Αμερικανοί έχουν κάνει τις επιλογές τους όσον αφορά αυτές τις άλλες δυνατότητες και εμείς στην Ευρώπη βεβαίως θα πρέπει να ξαναδούμε τις πηγές προμήθειας υδροκαυσίμων. Αν η Επιτροπή ζητάει συζήτηση για το θέμα, ας το συνεχίσουμε. Η γεωπολιτική της ενέργειας αλλάζει, εμφανίζονται νέοι παραγωγοί και πορεί όπως το συστολιθικό φυσικό αέριο, κατανέμονται πιο ισότιμα, διαφοροποιούνται περισσότερο και κυκλοφορούν σε περισσότερες αγορές. Σύντομα θα εκδημοκρατιστεί περισσότερο η ενέργεια, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό. Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης δεν είναι εγγυημένη. Πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε στο μεταλλασσόμενο ενεργειακό τοπίο το σχιστολιθικό φυσικό αέριο χάρη στην επανάσταση μπορεί να παίξει πολύ πιο μακροπρόθεσμο και σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα από ό,τι θεωρεί η Κομισιόν στον ενεργειακό δικό της χάρτη και να επιτρέψει μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών. Επίσης, οι υπεραισιόδοξες υποθέσεις της Κομισιόν όσον αφορά την επίτευξη των διαπραγματευμένων στόχων θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σενάριο β σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Πρέπει να ενισχύσουμε την αναμενόμενη ενεργειακή πολιτική. Έχουμε εργαλεία, αγορά, ανταγωνισμό, τις συνθήκες, την ενεργειακή πολιτική. Θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και να φροντίσουμε να συντονίσουμε τις αγορές ενέργειας και εκτός Ευρώπης και εκτός Ένωσης και να πραγματοποιήσουμε και κοινή αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τζόρνταν. Ένα λεπτό κυρία Τζόρνταν, συγγνώμη, το βιώσιμο ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι σήμερα. Θα υπάρχουν περισσότερες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και το μερίδιο των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα αλλάξει τα σημερινά τεχνικά χαρακτηριστικά ολόκληρου του σημερινού ηλεκτρικού συστήματος. Αυτό σημαίνει αλλαγή του συστήματος παρά των σχεδίων. Το σύστημα θα είναι πιο αποκεντρωμένο και πιο ευέλικτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι απλά Πρέπει να αναπτύξουμε έξυπνα δίκτυα smart grids. Χρειαζόμαστε επίσης και μια δυναμική παραγωγή ε, αποθεμάτων ενέργειας. Θα χρειαστούν τεράστιες επενδύσεις και τα δημόσια κονδύλια θα είναι μόνο η αρχή. Επειδή ο προπολογισμό είναι πολύ περιορισμένος. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα ικανοποιητικό επενδυτικό περιβάλλον με υποσχέσεις σταθερότητας. Έτσι λοιπόν εγώ προσωπικά υποστηρίζω νομικά δεσμευτικούς στόχους μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 και πάλι κάνω έκκληση στην Κομισιόν να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια που θα επιτρέψουν τη δυνατότητα να επιτευχθούν ε, στόχοι που, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν από τις παγκόσμιες συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, συνεργασία της, για την ατμόσφαιρα στην οποία προτιμάστηκε η έκθεση αυτά που είπαν οι Ευρωπαίοι, από, την, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικά. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια μακρά προοπτική και αυτό είναι σημαντικό και για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές. Ωστόσο, ο αριθμός των τροπολογιών και όλα τα διαφορετικά σενάρια που ενέχονται έχουν παραφορτώσει το κείμενο, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό, αν θέλετε, σε πολλές ε, περιπτώσεις των ε, εκθέσεων του Κοινοβουλίου. Άρα όλοι ζητούν κάτι για τον εαυτό τους σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια, σε ό,τι αφορά την ενέργεια από άνθρακα. Πρόκειται για το σωστό μείγμα, αλλά οι αποφάσεις που θα σήμερα θα επηρεάσουν το μέλλον και πολύ φοβόμαστε ότι σήμερα α, έχουμε προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να τα απεξέλθουμε και να απορριθούμε και δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων αυτή η έκθεση. Αφενός έχουμε ανεξέλεκτες επενδύσεις στη Γερμανία σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο σημαίνει ότι πολλές, πολλά εργοστάσια παραγωγής αερίου θα αποχαρακτηριστούν. Έχουμε κοινού κανόνες σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να καταστεί όμως μια πραγματικά κοινοτική αγορά αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόιλ, δύο λεπτά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την κυρία Τζαβέλα, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστη η συνεργασία μας. Στο θέμα αυτό, Ε, βλέπουμε έναν διαφορετικό τρόπο διεξαγωγή πολιτική συζήτηση. Και αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλα το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα υποβάλλει διαφορετικά σενάρια και μα καλεί να σκεφτούμε τι θα σημαίνει η απόφαση ΑΒΓ. Ίσως αυτό να συνέβαλε στο ότι θεωρούμε ότι είμαστε προειδοποιημένοι πλέον σε ό,τι αφορά ε, συμφωνία για νέα αριθμητικά στοιχεία. Αυτό όμω που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε μια αντικειμενική συζήτηση βάσει των σενάριων αυτών. Δεν πρόκειται για το τέλος μιας διαδικασία, ίσως για ένα σημαντικό βήμα να πρόκειται. Να μην θέσουμε πάντα μια πλειάδα στόχων, αλλά να κοιτάμε αντικειμενικά μεμονωμένα ε, στοιχεία. Και Θεωρώ ότι είναι σωστό το γεγονό ότι κοιτάζουμε όλε τι εναλλακτικέ λύσει. και, και ότι κοιτάμε και τα θέματα σχεστολιθικού αερίου και το πώ θα μπορούσε στο μέλλον να παράγει ενέργεια. Κατά πόσον ε, η ενέργειά μα είναι στι σωστέ τιμέ, τι αντικτύπωση υπάρχει στο περιβάλλον. Όλα αυτά δεν μπορούν να οριστούν από ένα μονομένο μεγάλο έργο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να τα κοιτάξουμε εγκάρσια όλα αυτά. Και άρα θεωρώ ότι είναι σωστό το ότι δείξαμε προσοχή για να μην ε, συμφωνήσουμε πάλι για νέα αριθμητικά στοιχεία, αλλά οι στόχοι όταν τίθενται να έχουν αλληλεπίδραση και με άλλους στόχους και θεωρώ ότι αυτό θα μας βοηθήσει να μην πετύχουμε το αντίθετο από τον στόχο μας. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει αυτό το ενδιάμεσο βήμα, που υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα, αλλά όχι το τέλος μιας διαδικασίας. Και ανυπομονώ να δω και το πράσινο βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής από τους σοσιαλιστές, ο κύριος, η κυρία Φαμπρέμπτε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντα την εισηγήτρια. Δεν είναι νομοθετικό το έργο, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική η έκθεση και το είπε και ο επίτροπο. Η εισηγήτρια πολύ δεσμευμένη ήταν και πάρα πολύ ε, επικοδομητικό πνεύμα έδειξε για να πετύχει αποτελέσματα. Φυσικά δεν ξέρουμε τι θα ισχύει το 2050. Κανείς δεν έχει ε, μαντικές ικανότητες, αλλά απεδείχθηκε από την προηγούμενη συζήτηση ότι τώρα θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια. Και εγώ σας το λέω, ε, το 2050 θα εξετάσω τι έχει επιτευχθεί. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα και την ομάδα μου και έτσι θα ψηφίσουμε αύριο είναι να μην κρυβόμαστε για πράγμα, πίσω από πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά να κάνουμε αυτά που πραγματικά πρέπει να κάνουμε, να, κάνουμε, να δώσουμε μια καλή προσέγγιση, να θέσουμε στόχους δεσμευτικού, να δούμε τους στόχους του 2020, το 2020, ε, να δούμε τι πετυχαίνουμε, τι δεν πετυχαίνουμε και μετά σε ό,τι αφορά το 2030 να θέσουμε νέους σαφεί στόχους σε ό,τι αφορά το 45% για παράδειγμα της 100 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και σε ό,τι αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και την ενεργειακή αποδοτικότητα. ο επίτροπο τα υποστήριξε αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και καλό λοιπόν του συναδέλφου προ τα δεξιά μα να τα υποστηρίξουν όλα αυτά αύριο για να αποστείλουμε ένα σαφέ μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, είναι πολύ ενδιαφέρον ο δικός χάρτη. Ε, ελπίζω να συμφωνήσετε και με τη γνωμοδότησή μα, αλλά δεν είστε πρόεδρος ε, ενός ε, think tank. Είστε πολιτικός ηθήνοντας και λοιπόν από τα πολιτικά σενάρια θα πρέπει να κάνετε μία επιλογή. Έχουμε και τις ε, no regret options. Τώρα λοιπόν θα πρέπει... Κλείνω πρόεδρε, κλείνω πρόεδρε. Βάσει αυτών των no regret options θα πρέπει να φροντίσουμε το 2050 να έχουμε πλήρη ανεξαρτησία στον τομέα τη ενέργεια, να εξαρτώμαστε μόνο από νέο Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θέλετε να απαντήσετε σε μπλε ε, κάρτα από τον κύριο Ρούμπιχ. Ο κύριο Ρούμπιχ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι η επιτυχής ιστορία της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τη μείωση των διοξιδίων του άνθρακα και των σχετικών αερίων ακολουθούμε το σχέδιο και νομίζω ότι μέχρι το 2020 η Ευρώπη θα είναι η πλέον υποδειγματική περιοχή όλου του κόσμου. Ρωτώ την κυρία Μπρέμπτ, πώς θα προχωρήσουμε. Μήπως αντί για το ETS θα έχουμε ένα cap and ε, prune fit σε ό,τι αφορά την παραγωγή με περιορισμένους ρήπους και να μειωθεί έτσι και ο ΦΠΑ για τους καταναλωτές και να είναι καταστούν πιο ενεργειακά αποδοτικά όλα αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση και με απασχολεί ιδιαίτερα και απασχολεί ιδιαίτερα και τη βιομηχανία. Θα πρέπει αυτά να τα ισορροπήσουμε. Είναι μια άλλα διαφορετική συζήτηση αυτή, αλλά είμαι πεπισμένη ότι το τρέχον σύστημα ανταλλαγής ρήπων δεν λειτουργεί και θα πρέπει να κοιτάξουμε το carbon footprint, αυτό το αποτύπωμα σε άνθρακα, προκειμένου να ξέρει ο καταναλωτής τα προϊόντα που αγοράζει, είτε είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, ε, έχουν την ίδια ποιότητα. Μόνο που αυτό, συνάδελφοι, προαπαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο και ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να περάσει το σύστημα ανταλλαγής ρηπών. Αν περάσουμε σε μια εναλλακτική λύση, Πρόεδρε, θεωρώ ότι σημαντικό είναι να υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε το ένα και να μην εφαρμόσουμε τίποτε άλλο, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε σημειώσει οποιαδήποτε πρόοδο. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ενδιαφέρουσα η βαλλοντική συζήτηση για θέματα αυτά. Σα Σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η μπλε κάρτα σημαίνει μισό λεπτό ερώτηση, μισό λεπτό απάντηση. Ο κύριο Τουρμές από την ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Τζαβέλα και από πλευράς του κυρίου Ζαντό, ο οποίος έκανε τις διαπραγματεύσεις από πλευράς των Πρασίνων. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς, ο Επιτρόπος έχει δίκιο που λέει ότι για το 2030 χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους για το κλίμα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προσέθετα και για την ενεργειακή αποδοτικότητα, γιατί η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι η μοναδική ρεαλιστική απάντηση στην ε, ενεργειακή ένδυα. Να μην αυταπατώμαστε. Η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου δεν καθορίζεται από εμά. Το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε του πολίτε να εγκαταλείψουν την θέρμανση με πετρέλαιο και να μπορέσουν οι το ε, αυτοκινητοβιομηχανίες να παράγουν αποτελεσματικά αυτοκίνητα για το αέριο. Κάποιοι πιστεύουν σε αυτό το θαύμα του συστολιστικού αερίου. Άμα ναι, είμαστε ρεαλιστές, καταρχάς είναι πάρα πολύ βλαβέ για το περιβάλλον. Κατά δεύτερον, το συστολιστικό αέριο στην Ευρώπη θα είναι δαπανηρή η παραγωγή. Να μην ε, ονειρευόμαστε τιμές όπως αυτές της Αμερικής. Αυτό πολύ απλά δεν είναι ρεαλιστικό και γι' αυτό λοιπόν έχει δίκιο η κυρία Γιόρταν που λέει ότι σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό θα πρέπει να αντικαταστήσουμε δύο τρίτα των εργοστασίων και σχεδόν όλο το δίκτυό μας. Αυτό πώς θα γίνει να επιτευχθεί με μια αυτήνη τιμή ηλεκτρισμού αν στους επένδυτες δεν δώσουμε κέρδη δεν θα επενδύσει κανεί. Και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικά για να περιορίσουμε και το κόστος. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω στη συζήτηση. Τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να είναι διαφανή και θα πρέπει να είναι και επίκαιρα. Το, το μοντέλο σας σήμερα έχει δύο σφάλματα να παρουσιάσει. Καταρχάς, δεν έχει παρουσιάσει ένα σενάριο υψηλής αποδοτικότητας και υψηλών ε, ε, ποσοστού ανανεώσιμων. Και κατά δεύτερον, το ατομικό κόστος είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Δηλαδή θα έπρεπε ίσως να κοιτάξετε και το κόστος το οποίο υπολογίζετε να αποτυπώνει το ρεαλιστικό κόστος. Ιδάλλως θα θέσουμε λάθος μηνύματα ως πολιτική. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας δώσουμε το λόγο για μισό λεπτό αν θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου Μπάστον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τούρμες, είμαι βέβαιος ότι πάρα πολύ σωστά ζητεί περισσότερη ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Όμω, εάν ήμασταν αρκετά τολμηροί τόσο να πάμε στην πράσινη ενέργεια από του ε, υδρογονάνθρακε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε χωρί να κλείσουμε τα φώτα ή χωρί να χρειαζόταν εξοικονόμηση ενέργεια. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα σωρό ηλιακή ενέργεια στην έρημο και να είχαμε την ίδια ενέργεια από στον κόσμο και τότε να είχαμε αρκετή ενέργεια από την αιωλική ενέργεια, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ε, διονύσουμε τι γεννήτριε. Οπότε αν όλα αυτά ήταν έτσι, τότε η αποτελεσματικότητα δεν θα ήταν τόσο σημαντική και τότε θα μπορούσαμε να καλύψουμε τι ανάγκε όλων. Παρακαλώ, απαντήσατε. Γκρέμπλε, κύριε Στουρμέ, έχει δίκιο. Έχουμε αρκετή ενέργεια και από τον άνεμο και από τον ήλιο. Όλο ο κόσμο μπορεί να έχει ενέργεια και γι' αυτό και πιστεύω ότι εσεί θα μπορέσει να συμφωνήσει με αυτό το οποίο θέλουμε, τόσο να έχουμε νέες ενέργεια παντού, αλλά ε, αποτελεσματικό σημαίνει έχουμε 100% σε χαμηλότερο κόστος ανανεώσιμα. Διότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι πάντοτε ε, το πιο ε, φθηνό από σε επενδύσεις και γι' αυτό και χρειαζόμαστε να υπάρχει αυτό το τρίγωνο ε, αποτελεσματικότητα, ανανεώσιμα και ευφύ δίκτυα. Και έτσι έχουμε επομένω το, το, το σύνδεσμο αυτό, τη σχέση, τη συνάφεια που λείπει. Ε, σας ευχαριστώ και τώρα πάμε στον επόμενο ομιλητή ο οποίος ε, θα μιλήσει για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και είναι ο κύριος Σιμάνσκι. Ε, σας ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση είναι κύμα πάρα πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων. Είναι ένα συμβασμό που κλείσαμε που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συναυθεί και δεν είμαι θα θέση να συμφωνήσουμε για την παράγραφο 91 και αυτό διότι κάνει ακόμα πιο σφιχτή την ε, πολιτική. Το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται ακόμα πιο μεγάλη δαπάνη για τη χημική βιομηχανία, για την ε, βιομηχανία παραγωγή χάρτου κλπ. Πρέπει να κάτσουμε να ανταγωνιστούμε με Ρωσία, με Αμερική, με Κίνα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μιλάμε για εισαγωγέ, μιλάμε για ε, διαπραγματεύσει ελευθερών εμπορίου. Επομένω, είναι επιστημονική φαντασία το να απαλλαγούμε από το διευθυντικό του άνθρακα. Και σύμφωνα με την ε, ε Ατομική Επιτροπή, την Διεθνή Επιτροπή μάλλον Ατομική ενέργεια, η περισσότερη ενέργεια θα προέλθει από κάποιε πηγέ που έχουν σχέση με ορυκτά. Επομένω, η σχετική δεσμενή διάκριση βάρο αυτών των πηγών δεν έχει μόνο δεν είναι αλλά και παραβλάπτει τον ενεργειακό μα τομέα και μα μπλοκάρει τι ε, επενδύσει και έτσι δεν έχουμε σταθερότητα και έτσι γίνεται η ενέργεια την οποία καταναλώνουμε πιο ακριβή σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρο. Και τώρα, από ό,τι μου λένε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Επομένω, δεν μπορώ να δεχθώ άλλε ε, μπλε κάρτες. Αλλά ο κύριο Ρώση έχει το λόγο και έχει το λόγο για 1,5. Δεχόμαστε την έκθεση της συναδέλφου. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πηγές ενέργειας και σε σχέση με τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα απόβλητα. Η συνάδελφος μιλάει για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας που θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 2014 με διαφάνεια τιμών λαμβάνοντας υπόψη και το περιβαλλοντικό κόστος και τους φόρους κατανάλωσης. Ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Μπούζεκ, είχε διοργανώσει συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς για να δημιουργηθεί αυτή η κοινή ε, ολοκληρωτική, ολοκληρωμένη πορεία ενέργειας. Κρίμα που δεν φτάνασαμε σε αίσιο πέρας. Θα ήθελα να πω ότι από πλευράς κόστους υπάρχουν διαφορές που είναι απαράδεκτες μεταξύ κρατών γιατί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία είναι πάνω από 130% της Γαλλίας ή της Πολωνίας και 80% πάνω από της Γερμανίας και 400% πάνω από το αμερικανικό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ ε, βιομηχανιών. Τη στιγμή που μιλάμε για τέτοιες διαφορές έχει μεγαλύτερη σημασία η μετεγκατάσταση. Προωθείται η μετεγκατάσταση. Ματίας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για τις ε, δύσκολες διαπραγματεύσεις. Η κυρία Τζαβέλα ξέρει ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρότασή της, ούτε εκείνη της Κομισιόν. Η πρόταση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τα κατά θέματα στον ενεργειακό τομέα του παρόντος. Όταν μιλάμε για ελάχιστους ε, πόρους και δεν έχουμε δεσμεύσεις ε, σαφείς ως προς τις ανανεώσιμες τη στιγμή που δεν λαμβάνουμε υπόψη την ενεργειακή απόδοση παρά μόνο για να τονώσουμε την οικονομία, Τη στιγμή λοιπόν που ενισχύουμε και τα πυρηνικά στην Ευρώπη, δύο χρόνια μετά την τραγωδία της Φουκουσίμα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, διότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία δυνατότητα στρατηγικής ευελιξίας. Περνάμε τώρα στους ανεξάρτητους ε, Σόζα Βάγνερ. Με βάση τον ορίζοντα 2050 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το μέλλον του Κοινοβουλίου μέσα στα πλαίσια ενός ε, προγραμματισμού. Γι' αυτό είναι επενεταίο το έργο της συναδέλφου όμως. Δεν ε, χειριστήκαμε πολύ καλά ορισμένα θέματα όπως τα ε, ορυκτά καύσιμα ή ανανεώσιμες, όπου υπάρχουν πολλά προσκόμματα που δημιουργούν σύγχυση στις επιχειρήσεις. Οι πολίτες όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να αποταμιεύουν ενέργεια και γι' αυτό δεν δεχόμαστε την κατασπατάληση ενέργειας που βλέπουμε σε πολλές πόλεις όπως σε αθλητικές εκδηλώσεις ή πανηγυρικές ε, εκδηλώσεις καθώς και την αποστολή μηνυμάτων μέσω δικτύων. Εάν δεν συγκρατηθούμε σήμερα, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι για αύριο. Στη συνέχεια, Καρίνς για δύο λεπτά. Κύριε Πίτροπε. Πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές που θα λάβουν υπόψη το επιχειρησιακό μας πνεύμα. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλάμε για ε, πράσινη ενέργεια μόνο και μόνο σαν να είναι αυτός σκοπός. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τρεις πτυχές. Καταρχήν, θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δεύτερον, θα πρέπει να μην είμαστε τόσο εξαρτώμενοι από εισαγωγές ενέργειας και θα πρέπει να έχουμε σταθερές τιμές που να είναι δίκαιες για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Αυτά μπορούμε να τα επιτύχουμε συνδυάζοντας διάφορες επιλογές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ανανεώσιμες, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να αποκλείουμε και την έρευνα για το σχιστολιθικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική πηγή για το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Της είπα, έχει μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση διότι ακριβώς χρησιμοποιείται σχιστολιθικό αέριο. Όσο περισσότερο παράγουμε, τόσο λιγότερο εισάγουμε και δεν αποκλείουμε και τη δυνατότητα να προωθήσουμε την πυρηνική ενέργεια. Ξέρουμε ότι ορισμένες χώρες είναι πολύ προηγμένες σε αυτό το τομέα, άλλες όχι και τόσο πολύ. Αλλά δεν είμαστε απομονωμένοι. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διάρθρωση τιμών, γι' αυτό θα πρέπει να εξισορροπήσουμε όλες αυτές τις πτυχές. Ε, Κυρία Μαντουρέλ, ευχαριστώ. Αυτός ο ενεργειακός χάρτης ε, προβαίνει σε μεγάλες αλλαγές. Μιλάμε για μείωση των ανθρακούχων εκπομπών. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τονώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Και επειδή θα πρέπει να έχουμε καθαρή ενέργεια, θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους ε, για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και θα μειωθεί η τιμή ενέργειας για τον καταναλωτή και η εξάρτησή μας από την αλλοδαπή. Όπως είπε και η κυρία Βαμπρέμ, υπάρχουν ορισμένα τμήματα της έκθεσης που θα πρέπει να αναλύσουμε περαιτέρω. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και να ορίσουμε υποχρεωτικούς στόχους. Επίσης θα πρέπει να προτρέψουμε την Επιτροπή να προωθήσει το καλύτερο δυνατό σενάριο για την βιωσιμότητα και την ενεργειακή μεγάλη σημασία για μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Χέλμαν. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Άριστα. Πάρα πολλά τόσα λέει. Βεβαίως θα έπρεπε να ασχοληθεί και με την αιμονή μα όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη μείωση των εκπομπών παρά το ότι εδώ και 17 χρόνια δεν έχει θερμανθεί το κλίμα. Παρά όλα αυτά, με χαρά μου βλέπω ότι τρέχουμε καινούργιε τεχνολογίε πρώτη εδώ πέρα, όπω α πούμε λιγνίτη, πυρηνική ενέργεια, ε, ε, ναι, α μείνει το φυσικό αέριο, μια που έχουμε την ευκαιρία που μα δίνει το ε, και να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές, τι θα γίνει με την φτώχεια την ενεργειακή. Η παράταξή μας δεν μπορεί να δεχθεί αυτά σχετικά με τις ανανεώσιμες διότι δεν είναι αποδοτικές πηγές ενέργειας, δεν είναι σε καλές τιμές. Θεωρούμε ότι όλα αυτά οδηγούν σε ναυάγια. Ούτε μπορούμε να συμφωνήσουμε με την αποθήκευση ε, του διοξιδίου και αυτό είναι άγριστο και κοστίζει πολύ και όσον αφορά αυτή την παγκόσμια δράση, τέτοια πράγματα είναι παραμύθια και αυτό επίσης ε, είναι ασύμφορο οικονομικά και δεν χρειάζεται και παρακαλώ συνάδελφοι ε, σας καλώ ε, να απόσχετε, έτσι σαν, σαν χειρονομία προς τη συγκίτρια, αλλά δεν μπορούμε να το επιψηφίσουμε. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκρίφιτ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, απόψε πολλές εκατοντάδες συνταξιούχων στη Βρετανία πρόκειται να πεθάνουν από το κρύο. Γιατί ακριβώ υπάρχει αυτή η παινία σε σχέση με το καύσιμο. Και οι βουλευτές θεώρησαν ότι αυτό το οποίο καταφέρνουν είναι ότι θα καταστραφεί ο κόσμος από την υπερθέρμανση. Αυτά δεν είναι κανένας είδους παραμύθι για το κατηχητικό. Αυτό είναι μια από τι πιο μεγάλε απάτε στην ανθρώπινη ιστορία. Όλα αυτά που λέμε για το διοξίδιο ε, ωφελούν κάποιου πλούσιου και ο κοινό άνθρωπο παγώνει. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι στόχοι δεν έχουν σχέση με τι ανάγκε του, του μέσου ανθρώπου, ο οποίο πεθαίνει κυριολεκτικά στο κρύο. Αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα είναι πρόκειται για ένα έγκλημα εκ μέρου των ε, μεγάλων εταιριών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα. Φτάσαμε στη διαδικασία Catch the Eye. Δώδεκα συναντούν στο λόγο. Ε, έξι από αυτού θα ικανοποιηθούν. Κύριο Σκέλη. Χαίρομαστε πάρα πολύ με τη στροφή που έχουν λάβει τα πράγματα με αυτή τη συζήτηση αλλά και με την προηγούμενη. Ευχαριστώ ιδίω την συγκεντρία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τόσο επόμενο ήταν πάρα πολύ λογικά και ξέρετε ότι θα πρέπει βέβαια η Ευρώπη να θεωρήσει ότι η ανταγωνιστικότητα είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Και επίση, εάν θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική Ευρώπη, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια ενέργεια που να είναι σε τιμέ συμφέρουσε. Θα πρέπει ομένω να φροντίσουμε έτσι και του ενεργειακού μα πόρου, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο τι υπάρχει, στο τι διατίθεται και βεβαίω θα ήθελα πάρα πολύ να έχω περισσότερες ομοιόμενες ενέργειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε τίποτα. Ε, γίνει λογική χρειάζεται. Να καταλάβει ότι η λύση είναι το energy mix, το μείγμα. Προσοχή, μην είμαστε δογματικοί. Συνεχώς βρίσκεται τεχνολογία. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για το πώς θα επιλύσουμε διάφορα θέματα τα οποία τώρα Μπορεί να είναι προβληματικά, αλλά ενδεχομένως στο μέλλον να είναι κάτι το λογικό, κάτι το θετικό. Πρόκειται για ένα εγχείρημα ελευθερίας. Έτσι μόνο μπορούμε να ορίσουμε το μέλλον. Μία μακροχρόνια πολιτική θα μας επιτρέψει να επιβληθούμε στην παγκόσμια αγορά της βιομηχανίας και της ενέργειας. Η Ευρώπη θα πρέπει να καταστεί πιο ανταγωνιστική. Η ενεργειακή πολιτική έχει μια κοινωνική διάσταση. Ορίζει και το μέλλον μας. Θα πρέπει να ορίσουμε δίκαιες τιμές προς τον καταναλωτή και να επινοήσουμε μηχανισμούς έλλειψης διακρίσεων. Ευχαριστώ. Köszönöm szépen τον ευχαριστώ. Ο κύριος Πασκάλ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Στην πρώτη δεκαετία του αιώνα μας οι ευρωπαϊκές χώρες έβγαλαν περίπου 200.000 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 2011 αυτό το ποσό έχει φτάσει το 488.000 δισεκατομμύρια ανά έτος. Ε, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε δει βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ούτε στη βιομηχανία, ούτε και στα νοικοκυριά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ε, εξαρτάται από τις εισαγωγές στον τομέα της ενέργειας και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κατανάλωση. Αποδέχομαι τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων σε 55% μέχρι το 2050. Πιστεύω ότι στην παρούσα φάση ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες ε, προβλέψεις, θα πρέπει να προβλέπουμε επαρκείς ε, ικανότητες βάσει όμως των δικών μας ε, ικανοτήτων. Ξέρουμε κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προβλέψεις. Αν θέλουμε να γίνουν οι μειώσεις μέχρι το 2050, θα πρέπει να γίνεται παραγωγή ενέργειας χωρίς διοξείδιο του άνθρακα Ξέρουμε ότι ένα θέμα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι άμα χαιρετίζουμε την πυρηνική παραγωγή πυρηνικής ενέργειας ως μια μορφή ενέργειας χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, αλλά είδαμε τι έγινε στην Φουκουσίμα. Ε, βάζουμε κάτω από το χαλί το ενδεχόμενο ενός ατυχήματο και δεν ατυχήματος και δεν λαμβάνουμε υπόψη τις συνέπειες. Μας ε, προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια Γίνονται τέτοιες εικασίες ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ματούλα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ορισμένους όρους που είναι σημαντικοί για την ενεργειακή μας ασφάλεια. Καταρχήν, ε, ρύθμιση του ενεργειακού καθεστώτος στα κράτη-μέλη που θα λάβει υπόψη την απελευθέρωση της, ε, των τιμών αγοράς και δεν θα επιτρέψει τον αποκλεισμό αγορών. Θα πρέπει να τονίσουμε την ενεργειακή απόδοση των περιφερειών πολύ περισσότερο στη Ρουμανία υπάρχουν ε, γεωθερμικές πηγές ενέργειας που δεν έχουν τύχη εκμετάλλευσης εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Θα ήθελα οι αρμόδιες εθνικές αρχές να ορίσουν καλύτερα αυτή την αγορά και να άρουν τα προσκόμματα για την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας καθώς και προώθηση των δικτύων μεταφοράς. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μειωμένο, ε, κόστος. Οι ανθρακούχες εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν και παράλληλα θα πρέπει να προωθήσουμε και το φυσικό αέριο ε, το οποίο έχει υγρή μορφή στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Ευχαριστώ. Άλβες. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ενωτική μας στρατηγικής για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Θα πρέπει να απαντήσουμε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πιο απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές γιατί βρίσκονται σε γεωγραφικό απομονατισμό. Θα ήθελα να ευαισθητοποιηθεί η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις για να μην επιλύουμε επιμέρους προβλήματα αλλά να διευρύνουμε το δίκτυο των ανανεώσιμων όπως ισχύει στις Αζόρες που έχουν ξεπεράσει και τους στόχους της Ένωσης για το 2020. Όμως, κύριε Επίτροπε, ε, δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις γι' αυτό. Αυτός ο δικός χάρτης θα πρέπει να επεκταθεί και μέχρι το 2050. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Επιτροπός έχει το λόγο για να συνοψίσει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρε, Κύριε βουλευτές, θα ήθελα να κάνω μια, κάποια περιορισμένα σχόλια για να σας απαντήσω στις ε, παρατηρήσεις σας. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ηλικιακή αποδοτικότητα. Με ανοιχτέ πόρτες ε, σας υποδεχόμαστε. Ήταν δι... σωστό το γεγονός ότι θέσαμε τον στόχο του 20% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Το χρονικό σημείο. Ποιο είναι το χρονικό σημείο το κατάλληλο για να θέσουμε τη νέο στόχο. Είμαι ανοιχτός σε νέε προτάσεις, αλλά γενικά θεωρώ ότι παρακολουθούμε κατά πόσον έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη τις υφιστάμενες οδηγίες. Θεωρούμε και περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα για το 2012 και το 2013. Και Θέλουμε να κοιτάξουμε και άλλα μέτρα όπως το labeling, το eco-design και μέτρα που έχουν λεφτεί στα κράτη-μέλη που δεν προβλέπονται από την οδηγία. Και μέχρι τα τέλη της θητείας μας θέλουμε να κάνουμε μία πρόβλεψη για το κατά πόσο η ταχύτητα των κρατών μελών είναι επαρκή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή δηλαδή των δεσμευτικών μέτρων προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο του 20% μέχρι το 2020 ή κατά πόσο χρειάζονται και άλλα μέτρα σε ό,τι αφορά το 2015 ενδεχομένως. Τότε θεωρώ ότι η χρονική στιγμή θα έχει φτάσει για ένα νέο στόχο ενεργειακό βάσει των αναλύσεων των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο της αποτελεσμότητας ε, της κοινή μας οδηγίας των εθνικών σχεδίων δράσης δηλαδή εγώ τίνω και κλείνω να δούμε το 2030 να τεθεί ως νέος ε, στόχος για δεσμευτικούς στόχους. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν κάτι φιλόδοξο και ρεαλιστικό για το σχιστολιστικό αέριο. Συμφωνούμε όλοι ότι το αέριο έχει ιδιαίτερη ε, σημασία και στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα και αυτό για τρεις λόγους. Το αέριο σε μεγάλο βαθμό διατίθεται πολύ περισσότερο από ότι το πετρέλαιο. Κατά δεύτερον, το αέριο είναι σαφώς πιο φιλικό προς το περιβάλλον και για την βιομηχανική επεξεργασία, αλλά και για τη θέρμανση, αλλά και για την παραγωγή ηλεκτρισμού, από ότι για παράδειγμα ο άνθρακας. Και τρίτος λόγος, το αέριο είναι πάρα πολύ ευέλικτο και ιδανικό δηλαδή για ανανεώσιμες ενέργειες. Δηλαδή όταν δεν έχουμε αέρα, δεν έχουμε ήλιο, έχουμε πολύ πιο εύκολα διαθέσιμο το αέριο για την παραγωγή θερμότητας. Έχουμε λοιπόν μια ευρωπαϊκή αγορά ε, παραγωγής αερίου 540 ε, κυβικά μέτρα ανά έτος ένα τρίτο της ε, κατανάλωσης αερίου είναι από δική μας ε, παραγωγή. Όλες οι προβλέψεις όμως για τη συμβατική παραγωγή αερίου στην Ευρώπη τι λένε ότι οι ποσότητες αυτές μέχρι το 2030-2035 θα έχουν εξαντληθεί. Και τότε λοιπόν ερωτώ τι θα κάνουμε. Θα έχουμε 100% εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία, από την Αφηγία, από την Αλγερία. Από την Ιγυρία, από το Κατάρ, από τον νότιο διάδρομο. Θέλουμε δηλαδή 100% εξάρτηση από εισαγωγές, γνωρίζοντας βέβαια ότι στην ε, Νιγηρία, στην Ακτική, στην Αλγερία επίσης υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, γνωρίζοντας ότι οι εργασιακές συνθήκες για την ε, παραγωγή στη Σιβηρία δεν είναι απαραίτητο πάρα πολύ ευνοϊκές. Και το βασικό θα είναι ότι εμείς θα έχουμε το αέριό μας και ότι η εξόριξη, ο τρόπος εξόριξης, ο τρόπος εργασίας θα είναι κάτι που δεν θα μας απασχολεί. Εγώ προτιμώ να έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Το περιβάλλον είναι σημαντικό. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτό που πήγε στραβά και που πήγε καλά στην Αμερική. γιατί μπορεί να είναι ασφαλές το φυσιολογικό αέριο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αποκλείεται. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι γεωλόγοι μιλούν για την προστασία των υδάτων, των πόσιμων υδάτων της φύσης και θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί το δυναμικό του αερίου. Θα πρέπει αυτό να είναι η κοινή ευρωπαϊκή μας φιλοδοξία. Η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες, ε, η Μεγάλη Βρετανία θα προηγηθούν όλοι αυτοί και μετά θα ακολουθήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας. Και αν ε, μιλάμε για 10%, για 15% του ενεργειακού μείγματος που χρειάζεται η Ευρώπη, αλλά με ίδια παραγωγή, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε την ανάλογη επιρροή των, στους Ρώσους σε ό,τι αφορά την ε, σύνδεση με την τιμή. Δηλαδή, με κάποια ποσότητα αερίου θα έχουμε κάποιες επιρροές. Και να σας πω από τη συζητήσεις μου με τη Μόσχα, το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει σε ό,τι αφορά το συστολιστικό αέριο. Και ίσως σε κάποια χρόνια και η Ουκρανία να είναι και παραγωγός συστολιστικού αερίου που θα εξαγάγει αέριο στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που συστήνω είναι ανοιχτό πνεύμα και ανοιχτή προσέγγιση. Δεν είμαι υπεραισιόδεξος. Θέλω να υπάρχει ανοιχτός χαρακτήρας, επιστημονικός χαρακτήρας με συγκεκριμένα τεκμήρια. Το θέμα των ενεργειακών τιμών τώρα. Η ανάγκη του πρέπει να το εξετάσουμε εις βάθος. Είναι καλό το γεγονός ε, το ότι συζητάμε τις ενεργειακές τιμές. Γιατί ο οικονομικός ε, παράγοντας είναι σημαντικός σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο καταναλωτής φυσικά είναι ευαισθητοποιημένος σε ό,τι αφορά τις υψηλές τιμές. Και αυτά ισχύουν και για τις μετακινήσεις αλλά και για τις θερμάνσεις. Αλλά μπορεί να έχουμε φτάσει στο άνατο σημείο της, ε, των ενεργειακών τιμών και η ενεργειακή ένδυα δεν είναι πλέον κάτι το ξένο. Υπάρχουν πολίτες που σε ό,τι αφορά τη θέρμανσή τους, τη βενζίνη τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και θα πρέπει να προσαρμοστούν οι κοινοφιλείς υπηρεσίε και θα πρέπει η ενέργεια να συγκαταλεχθεί ε, όλο και πιο πολύ στο βασικό καλάθι βασικών αναγκών. Δεν ε, υποστηρίζω τις ε, επηρεασμένες τιμές. Θα πρέπει να ισχύσουν οι τιμές της αγοράς. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε και να λειτουργεί όχι μόνο η χοντρική αγορά, αλλά και η λιανική αγορά. Σε 20 κράτη-μέλη ακόμη οι καταναλωτές έχουν ρυθμιζόμενες τιμές που δεν αντιπακρίνονται στην προσφορά και στη ζήτηση και στην Ισπανία έχουμε το εξής πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά αυτές τις ρυθμιζόμενες τιμές δεν ακολουθούν τις ε, τρέχουσες ανάγκες σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να προωθούμε τις ανανεώσιμες, θέλουμε να προωθηθούν και ποτέ δεν ε, ασκήσαμε αντίθετη πίεση. Τελευταίο θέμα τώρα σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα 2020. Το θέμα των τεχνολογιών αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το, το θέμα της ποιότητας των ε, ε, δικτύων ε, παροχής ηλεκτρισμού πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα προσθεθεί και θέματα υγειοθερμικής. Ήμουνα την προηγούμενη Πέμπτη στην Ισλανδία και βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες πρόοδε στον τομέα αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταία η Νίκη Τσαβέλα, η συγγετριά μας, θα λάβει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, μου άρεσε η τοποθέτησή σας για την πολιτική των Ευρωπαίων να σταματάμε τις εξορίξεις αλλά να μην δίνουμε σημασία πώς γίνονται αυτές στις χώρες από τις οποίες εισάγουμε. Στην Αμερική αυτή την πολιτική των Ευρωπαίων την αποκαλούν «not in my backyard». Και μου άρεσε πολύ που το τοποθετήσατε. Κυρίες και κύριοι, στην έκθεση προσπάθησα να συμπεριλάβω τουλάχιστον όλες τις συγκλίνουσες απόψεις με μία μέση οδό έκφρασης. Γι' αυτό ήρθαμε και ε, ε, βγάλαμε ένα πολύ μεγάλο κείμενο θα έλεγα Όσον αφορά την ε, ενεργειακή εξοικονόμηση, ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Η έκθεση ε, εισηγείται το συγκεκριμένο θέμα να εισαχθεί στα προγράμματα εθνικής εκπαίδευσης ώστε η εξοικονόμηση ενέργειας να ξεκινάει από τις ρίζες, από το grassroots. Κύριε Επίτροπε, προσβλέπουμε με την έκθεση αυτή για μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για την ενεργειακή πολιτική από την Επιτροπή μέχρι το 2030. Μία έκθεση της Επιτροπής που θα ξεκαθαρίζει δεσμευτικούς στόχους, απλούς στόχους και την τύχη και το μέλλον των μορφών ενέργειας στην Ευρώπη. Έτσι θα ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι επενδυτές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τον οδικό χάρτη με τον οποίο θα πορευτούν στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Σας ευχαριστώ κυρία Τζαβέλα και ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Το επόμενο θέμα έχουμε την αξιολόγηση των κινδύνων και της ασφάλειας των